Good morning, dear colleagues. If Παρακαλώ καθίστε για να αρχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που επιτέλους με προσέξατε. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω ένα νέο μέλος της Επιτροπής μας, τον κύριο Ρούπερτ Μάθιους, σας ε, καλωσορίζουμε. Ο κύριος Μάθιους αντικαθιστά τον κύριο Ντάνκαν. Στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχουμε την υποβολή έκθεση σχετικά με τις τρέχουσες ε, διοργανικές ε, διαπραγματεύσεις. Είχαμε έναν τριμερή διάλογο σε σχέση με το πακέτο των αποβλήτων και μιλήσαμε για προετοιμασία σε τεχνικό επίπεδο το Συμβούλιο συνεχίζει να απορρίπτει τα, τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025-2030 σε σχέση με τα απόβλητα στον τομέα των τροφίμων και στο δεύτερο τμήμα του τριμερούς διαλόγου έγινε μία συζήτηση σε σχέση με τους στόχους και μέθοδο υπολογισμού εξαιρέσεις και ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις εν ώψη του τρίτου τριμερούς διαλόγου που προγραμματίζεται για τις 26 Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο θέμα είναι το ETS, ανταλλαγή εκπομπών. Είχαμε τον δεύτερο άτυπο τριμερή διάλογο σε σχέση με τη δική μας ε, θέση της 15ης Φεβρουαρίου και της εντολής της ΚΟΡΕΠΕΡ του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου. Τα τρία θεσμικά όργανα έλαβαν γνώση την, ε, τα μέτρα σε σχέση με την καλύτερη ευθυγράμμιση και παραγωγή ε, benchmarks και ποιοτικές αποτιμήσεις σε σχέση με τις ρυθμίσεις των τομέα των διαρών. Η Προεδρία συμφώνησε να παρουσιάσει συμβασμού στα κράτη-μέλη και μετά εκπροσωπήθηκε και η θέση του Συμβουλίου σε σχέση με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στον τομέα της αεροπλοείας ε, και της ναυσιπλοείας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα μέτρα που υπάρχουν με βάση το Ταμείο Μετάβασης. Υπάρχει και το λεγόμενο τρίγωνο ζητημάτων σε σχέση με τις ε, διαρροές άνθρακα και μιλήσαμε και για τους σχετικούς πόρους. Συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι θα επιτελεστεί πρόοδος ως προς το άρθρο 10D και τις διατάξεις MSR. Χτες έγινε ο τρίτος ε, τριμερής διάλογος όπου μιλήσαμε για τις μεταβλητές του Ταμείου και τα συναφή ζητήματα για να γίνει πρόοδος. Μιλήσαμε για την φιλοδοξία της πρότασης, ιδιαίτερα ως προς τις διατάξεις MSR και τα στοιχεία αναθεώρησης. Ζητήσαμε περαιτέρω επεξηγήσεις ως προς το σύνδεσμο μεταξύ benchmarks και, ε, ελεύθερες, και την ελεύθερη διάθεση ποσοστώσεων καθώς και διασταυρούμενα στοιχεία. Η ε, διπλή αυτή προσέγγιση αφορά και τις αποζημιώσεις. Επίσης, δυνάμει του άρθρου 10 Δέλτα συζητήσαμε τις εξαιρέσεις καθώς και τις επιδοτήσεις της τρίτης φάσης. Μιλήσαμε για τις ε, νέες διατάξεις του MSR στις 13 Σεπτεμβρίου προβλέπεται ο επόμενος ε, τριμερής ε, διάλογος και στο μεταξύ προβλέπονται δύο τεχνικές συναντήσεις. Ως προς το ΡΟΣ, στις 21 Ιουνίου είχαμε τριμερή διάλογο όπου φτάσαμε σε μια συνολική συμφωνία όπου ε, η δευτερογενής αγορά καλύπτει την ηλεκτρική και ηλεκτρονική αγορά μέσω ορός, καθώς και τα εξαρτήματα εάν τεθούν στην ε, αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2019. Σε σχέση με τα εξαρτήματα του ηλεκτρικού ηλεκτρονικού μηχανισμού θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα επιστροφών business to business. Επιπλέον η Επιτροπή θα πρέπει να χορηγήσει στους ετούντες τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα χρονοδιάγραμμα για την έγκριση των αποφάσεων ως προς τις εξαιρέσεις που θα υπάρχουν στους περιορισμούς ε, ως προς τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό μηχανισμό. Ο μηχανισμός εγκρίθηκε στις 28 Ιουνίου από την ΚΟΡΕΠΕΡ. Εμείς θα ψηφίσουμε τώρα το πρωί και στην Ολομέλεια θα συζητηθεί στην πρώτη σύνοδο του Οκτωβρίου το θέμα. Έχουμε και τη συμμετοχή των συναδέλφων. Στην 71η ε, συνάντηση του Διεθνής Οργανισμού Ναυσιπλοείας μέσα στα πλαίσια της προστασίας ΜΕΡΞΕ 71 θα υπάρξει αποστολή. η κύριοι Φαρία και Έικχαουτ ήταν παρόντες και θα ήθελα να μας πούν πώς, πώς έλαβε χώρα αυτή η αποστολή. Ο κύριος Φαρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ξέρετε είναι η τρίτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει μια αποστολή στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Ήταν η 71η Σύνοδος της Επιτροπής ε, Προστασίας ε, της, ε, του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, MEPC, και ήμασταν από τις 3 μέχρι τις 5 Ιουλίου, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, πριν από την συνάντηση που, έγι, που γίνεται ανάμεσα στις συνόδους. Ε, από τους πράσινους που εγώ και ο κ. Μπαζέκα, Και είναι η τρίτη φορά που η Επιτροπή ΕΜΒΗ στέλνει εκπροσώπους ε, στην MEPC. Ήταν η πρώτη φορά που συνεδρίασε η ομάδα εργασίας που συνεδριάζει μεταξύ των ε, συνόδων και η MEPC 71 ε, συζήτησε διάφορα θέματα καθώς και το όραμα, το επίπεδο φιλοδοξίας, κατευθυντήριες γραμμές, πρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα μέτρα και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη. Ήταν πολύ επικοδομητικέ συζητήσεις, όμως αν το θέμα είναι τι επετεύχθη ε, απτά συγκεκριμένα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η απάντηση είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση, ως συνήθω. Εμεί είχαμε την προστοκία ότι θα μπορούσαμε να είχαμε μια πολιτική δέσμευση, να συμφωνήσουμε πάνω σε παγκόσμιους τομεακούς στόχους μέχρι το 2018. Στο τέλος όμως των δύο εβδομάδων δεν υπήρξε τέτοια πολιτική δέσμευση. Μια άλλη προσδοκία ήταν να υπάρξει μια πολιτική δέσμευση να εφαρμόσουμε ε, προ, ε, βραχυπρόθεσμα μέτρα, το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχει ένα κατάλογο των μέτρων, καταρχά ε, διαχείριση τη ταχύτητα των πλοίων, ε, καθώ και πιο αυστηρά πρότυπα για το σχεδιασμό των πλοίων. Όμω, είναι απλώς ένας κατάλογος αυτός, δεν έχουμε καμία δέσμευση ότι θα συμφωνήσουμε και πιο σημαντικό ότι θα εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα ε, το συντομότερο δυνατόν. Αυτό όμως θα ήταν πολύ ε, σημαντικό, ούτω ώστε να ασχοληθούμε με τι εκπομπές των πλοίων για να υλοποιήσουμε τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με την αναμονή και να συζητάμε απλώς. Ε, υπήρξαν και κάποιες αρνητικές ε, εξελίξεις ε, στην MEPC 71. Ε, στις αρχές του επόμενου χρόνου δεν θα συζητήσουμε την, τα πρότυπα για τα νέα πλοία και ε, τις αρχές του 18. Καθυστερούμε μέχρι το 19. Επομένως, τα πλοία που σχεδιάζονται σήμερα θα, θα συνεχίσουν να πουλούνται. Ε, όμως οι τομεακές εκπομπές ε, θα πρέπει να μειωθούν δραματικά αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις καθυστερήσεις. Μία άλλη αρνητική εξέλιξη ήταν ότι ο IMO αποφάσισε να μην ε, ε, έχει πρότυπα για τον τρόπο συλλογής δεδομένων δεν υπάρχει κανένα, καμία διαφάνεια και πόρα απέχει το σύστημα του IMO από το ανοιχτό, διαφανές και στεναρό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης δεν ξέρουμε θα γίνει με το κανονισμό παρακολούθησης ε, για την παρακολούθηση, την αναφορά και την επαλήθευση, το MRV. Επίσης, ε, η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση το δικό μας CTS είναι ότι θα πάρουμε μέτρα ε, μόνο αν δεν υπάρχει συγκρίσιμο σύστημα ε, στα πλαίσια του IMO. Αυτές τις δύο εβδομάδες μοιάζει ότι ο ναυτιλιακός τομέα θα συμπεριληφθεί στο νέο ETS. Ε, e ο IMO συνεχίζει να κάνει πολλές συνεδριάσεις, πολλές διμερείς συνεδριάσεις, ε, πολλά ευχολόγια, πολλά λόγια, αλλά πολύ λίγα από τα αποτελέσματα. Εγώ πιστεύω ότι το να αποτύχουμε δεν είναι επιλογή. Η αναμονή δεν είναι επιλογή. Αυτά είναι τα συμπεράσματα μετά την τελευταία συνάντηση της περασμένης εβδομάδας, καθώς και της ε, Intersessional, ε, δηλαδή της, ε, συνα, της μεταξύ των δύο, της συνεδρίασης μάλλον μεταξύ των δύο συνόδων, που ήταν την, προ την προηγούμενη από την, ε, την προ προηγούμενη συγγνώμη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν ο Μπάς θέλει να σχολιάσει. Ας περιμένουμε την επόμενη MEPC και όπως λέμε και στη χώρα μου, Ινσαλά. Μακάρι να τα καταφέρει η MEPC, δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Ευχαριστούμε κύριε Φαρία. Ο κύριος Έικχαουτ, ο άλλος πυλώνας αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με δίνετε το λόγο για να πούμε τι έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο στην Σύνοδο του Διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού. Ήταν μεγάλη αποστολή δύο ατόμων και ο κύριος Γιούνκερ ε, δυσαρεστήθηκε που δεν ήμασταν στην Ολομέλεια την τρίτη το πρωί και μέσα στο Λονδίνο. Μια κλασική συνεδρίαση του IMO που μπορεί να πει κανείς ότι το ποτήρι είναι μισοάδιο, μισογεμάτο ανάλογα με το πώ το βλέπεις. Αν προέρχεσαι από μέσα από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και έχει συνηθίσει στο ρυθμό των αλλαγών μέσα στον οργανισμό, ε, μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει μια αλλαγή διάθεση ε, λόγω των ε, νήσων του Ειρηνικού. Νησιά του Ειρηνικού όπως το Τουβαλού, τα νησιά Μάρσαλ, ε, φέρνουν ε, περισσότερο πολιτικό επίπεδο στην επιφάνεια, γιατί μέχρι τώρα είχαμε πιο τεχνικό επίπεδο με τα νεολόγια των πλοίων κλπ. Ενώ τώρα τα νησιά αυτά που έχουν καταλάβει την επίπτωση των κλιματικών αλλαγών ξέρουν ότι κάτι πρέπει να γίνει και γι' αυτό φέρνουν μια καινούργια δυναμική και αυτό είναι θετικό. Και από πλευρά IMO, τρίτη φορά πήγα εγώ εκεί, ε, βλέπει ότι υπάρχουν σοβαρέ συζητήσει ότι κάτι πρέπει να γίνει για την αλλαγή του κλίματο. Βέβαια, αν το δει κανεί από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι το εξή. Αποφασίστηκε ότι θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε μια στρατηγική που θα ε, υιοθετηθεί το 2018 και θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2023. Λίγο πολύ εκεί βρισκόμαστε ε, στον IMO. Η στρατηγική που θα υιοθετηθεί του χρόνου είναι σημαντικό να έχει ένα όραμα, να έχει στόχους, να έχει ε, τρόπους μέτρησης και να έχει βραχυπρόθεσμου μετρήσιμους στόχους και να μην περιμένουμε μέχρι το 2023. Και βέβαια θα έχει και μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Ξέρουμε ότι κάποια μέρη θέλουν να το προωθήσουν, ξέρουμε ότι τα νησιά του Ειρηνικού μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τη δύναμη να σπρώξουν κάποιες αλλαγές, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν είναι έτοιμες ακόμη να αναλάβουν δράσεις. Τέλη Οκτωβρίου και λίγο πριν από την ε, επόμενη ε, σύνοδο, την MEPC 72, έχουμε δύο ενδιάμεσες συνεδριάσεις και θα είναι κέρια σημασία να γίνουν οι συζητήσεις για να δούμε αν θα υιοθετηθεί αυτή η στρατηγική στην επόμενη σύνοδο, την 72η. Ο ρυθμός αλλαγών είναι πολύ αργός ακόμη. Αλλά ας δούμε τι μπορεί να γίνει γιατί έχουμε ακόμη ένα χρόνο μπροστά μας. Ας ελπίσουμε ότι η στρατηγική αυτή θα έχει και άμεσες δράσεις γιατί δεν μπορούμε ε, να περιμένουμε για υλοποίηση μετά το 2023. Τώρα, κάτι άλλο για το σύστημα συλλογή δεδομένων. όντω υπάρχουν πρόοδοι. όπω είπε ο κ. Φαρή, υπάρχουν μεγάλε διαφορέ με την ευρωπαϊκή προσέγγιση για το MRV, ιδίω για την διαφάνεια και την επαλήθευση από τρίτου, Και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να κρατήσουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Βεβαίω και να συζητήσουμε πώ θα ευθυγραμμίσουμε την ευρωπαϊκή προσέγγιση με την απόφαση του IMO, αλλά θα πρέπει να το δούμε ήταν πολύ χρήσιμη η παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σύνοδο αυτή. Η πολιτική πίεση αποτελεί ένα παράγοντα που κινητοποιεί τα συμβαλόμενα μέρη. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες για να επιταχύνουμε και τις αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. πρόεδρος των νησιών Μάρσελ ε, είχε παρευρεθεί σε μία συνάντηση ε, δική μας στο Στρασβούργο την τελευταία φορά. Έχουμε και εμείς λοιπόν κάπως μια άμεση παρακολούθηση. Η Επιτροπή νομίζω ότι θέλει να, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μιλήσει. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλω να, καλώς, καλημερίσω τα μέλη της Επιτροπής και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρευρεθήκατε το Λονδίνο, στη σύνοδο αυτή και που μας βοηθήσατε στις προσπάθειές μας να κινητοποιήσουμε τις άλλες πλευρές ε, για τα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν. Ήταν κέρια η συνάντηση αυτή στο να προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε τις περισσότερο διστακτικές αντιπροσωπείες. Συμφωνώ με αυτά τα οποία ελέγχθησαν ότι αρχίζει κάπως η στάση να αλλάζει. Αρχίζουν να αναγνωρίζουν το ότι πρόκειται για ένα οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών όπου συνενώνονται 173 κράτη που έχουν ναυτιλία με βάση τις συνενετικές διαδικασίες. Εξορισμού λοιπόν είναι πιο αργή η πρόοδος από ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού εκεί κινούνται με συνένεση και είναι τόσο περισσότερες χώρες, αλλά είναι θετικό το να δούμε ότι μια ομάδα χωρών που παραδοσιακά ε, μπλόκαραν τα πάντα όσον αφορά τη μείωση εκπομπών, ε, έχει αρχίσει να αναγνωρίζει τα προβλήματα και αρχίζει να υπάρχει πρόοδος. Η αξιολόγηση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι μέχρι το 2018 θα έχουμε μια αρχική στρατηγική. Συμφωνώ ότι θα χρειαστεί μέχρι το 2023 να περιμένουμε για να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, αλλά θέλω επίσης να πω ότι ο Διεθνής Δαυτιλιακός Οργανισμός ήταν ο πρώτος διεθνής οργανισμός ε, που κατέληξε σε υποχρεωτικά πρότυπα για ενεργειακά αποδοτικά σκάφη για το 2013 και αυτά τα μέτρα θα βελτιωθούν σιγά σιγά. Επίσης, όπως έγινε και για τη συλλογή δεδομένων, ό,τι αποφασίζεται από αυτόν τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να παίρνει κάποιο χρόνο, αλλά στη συνέχεια η υλοποίηση προχωρεί με γοργά βήματα. Θέλω επίσης να αναφέρω ότι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αύξηση δυνατοτήτων, χρηματοδότηση που δόθηκε ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ για την δημιουργία κέντρων συνεργασίας για την ναυτιλιακή τεχνολογία, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αναγνωρίστηκε από τις χώρες που ήταν πριν διστακτικές και ελπίζουμε ότι ε, θα μπορέσουμε στο μέλλον να επαυξήσουμε ε, ε, αυτή την προσπάθεια και στις διαπραγματεύσεις θα μας βοηθήσει η επιτυχία αυτού του έργου. Θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο που παρακολούθησε το σύστημα συλλογής δεδομένων για ε, να πει δύο λόγια για το πώς πιστεύουμε ότι από εδώ και πέρα θα προχωρήσουμε τα πράγματα. Ως προς το σύστημα συλλογής δεδομένων που ενέκρινε το MPC πέρσι το φθινόπωρο τον Οκτώβριο, θα ήθελα να πω ότι ενεκρίθησαν οι δύο τελικές κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την διαχείριση της βάσης δεδομένων και εδώ είδαμε ότι είχαμε θετική έκβαση της αξιολόγησης και η γραμματεία του IMO θα συμπληρώσει αυτά τα στοιχεία. Η δεύτερη κατευθυντήρια γραμμή αφορά την επαλήθευση των ε, στοιχείων που συλλέγονται και όπως ανέφεραν τα μέλη, εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ του ευρωπαϊκού και του συστήματος του IMO η αξιολόγηση, η επαλήθευση του IMO είναι πολύ υψηλότερων ποιοτικών προδιαγραφών. Το επόμενο ε, βήμα ε, για την Κομισιόν είναι η ε, αναθεώρηση του κανονισμού. Τώρα έχουμε ετοιμάσει την, από, την, τις επιπτώσεις, την ε, αξιολόγηση των επιπτώσεων και θα περάσουμε στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης. Ωραία, σας ευχαριστώ. Άρα ολοκληρώνεται το πρώτο τμήμα της ημερήσιας διάταξης. Περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε την ηλεκτρονική σας ε, κάρτα, να είσαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία. Έτοιμοι, ωραία. Ε, αρχίζουμε με τα εύκολα, από τα εύκολα. Έχουμε μία ενιαία ψηφοφορία για την αντίρρηση σύμφωνα με τη γενετικό τροποποιημένη σόγια. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η δεύτερη είναι για το ε, κείμενο που ενέκρινε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ονομαστική άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Έκθεση Γκάμπους. Διαδικαστική κανόνες στον τομέα των περιφαλλοντικών εκθέσεων. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά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 ψηφίσουμε για την απόφαση διαθεσμικών διαπραγματεύσεων. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Και εγκρίνεται. Να σας συγχαρούμε και ευχαριστούμε πολύ. Έκθεση Φλάναγκεν. Μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που δρούν στα του δημοσίου συμφέροντος. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Ε, θέλετε να ελέγξουμε, πολύ ευχαρίστως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Ελέγχουμε γιατί 40 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Το δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. πέρας εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε την 87. Ωραία, ελέγχουμε για την 87. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Για μία ψήφο. 88 υπέρ. 88 υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ,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 αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται. Πέρας και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. έκθεση Γκέρλιν ε, περιορισμοί προς τις αεροπλοϊκές δραστηριότητες. Βάσμος 1. Υπέρ. Κατά. Υιοθετείτε. Συμβάσμος 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 12. Όχι, τις ψηφίσαμε μαζί 11 και 12. Συμβιβασμός 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Τραν 10 και τροπολογία 90 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Ήτρε 13 υπέρ. Όχι, καταπί... καταπίπτει αυτή. Τροπολογία 17 υπέρ. Και αυτή καταπίπτει. Τροπολογία 91. Αυτή παραμένει. Υπέρ. Ναι, ναι, είπα, παραμένει. Την ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική λύση 6 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Μετά από πολλές σελίδες που Πάμε στην 125. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τραν 12. Υπέρ. Κατά. Ως ζητώ συγγνώμη. Πολλά χρώματα έχει αυτός ο κατάλογος. Συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. η 1 υπέρ κατά άποχες την ελέγχουμε χρονικά. Την ίτρε 1. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας προφορίας. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ίτρε 2. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 3 υπέρ κατά αποχές το ελέγχουμε. Δηλαδή την Ήτρε 3. Ηλεκτρονικά. Πέρας φοφορίας. Υιοθετείτε. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία ένα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Συμβασμός 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 42 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές αϊοθετείται. Σαράντα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 8 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τραν 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Και πάμε στην 52 υπέρ. Κα, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 55 υπέρ Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 6 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 10. Επίδειξα τίποτα. Όχι, ήτρε 10 υπέρ κατά αποχές. Δεν ξέρω τι κάνουν οι σοσιαλιστές. Είσαστε υπέρ ή κατά. Τότε υιοθετείτε. Θέλετε να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ναι, ελέγχουμε την ΙΤΡΕ 10 ηλεκτρονικά. Πέρας φοφορίας, υιοθετείτε. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Στα πέντε. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας της ψηφοφορίας και υιοθετείτε. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για το επόμενο που είναι έτσι παχουλό-παχουλό το κείμενο. Η επόμενη ψηφοφορία αφορά τη Λουλουσιεύ. Ξεκινάμε με την τροπολογία 94 υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Την 101 παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 134 τμήμα δεύτερο. Μαζί με την Άγκρη 21 τμήμα δεύτερο. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Για την 138 να ψηφίσουμε. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 147. Θέλετε να ελέγξουμε την 148 με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Όπως το είχαμε πει. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απολύπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ή να το ελέγξουμε την 159 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Αγκρί 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 162 όχι, καταπίπτει. Φτάνουμε στη συμβαστική 16α. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ή να ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τη συμβαστική τροπολογία 16α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 16β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η Ειτρια32. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η Ειτρια33. Υπέρ, κατά, Αποχές. Δεν είμαι σίγουρη. Οι σοσιαλιστές είναι υπέρ ή κατά. Δεν είναι σίγουρο. Ας το ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την ΙΤΡΕ 33 ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κύριε Λίντς. Είπαμε συμβαστική τροπολογία 5. Σελίδα 17 στη δική μου σελίδοποίηση, λέει η Πρόεδρος. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.48 2.47 συγγνώμη και Άγκρη 41 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.50 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Την 250 με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 251-252 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 254 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήτρε 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήτρε 39 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ή 40 υπέρ, κατά, αποχές, όχι, περάσαμε τη συμβαστική τροπολογία 12. Ψήφι υπέρ για την 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα φτάνουμε στην Ήτρε 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ή 42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρη 53 στη σελίδα 22 του καταλόγου μου. Ψήφι υπέρ για το, την Άγκρι 53 κατά αποχές απορρίπτεται. 2.92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 1 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την Ήτρε 1. Άρχεται η ψηφοφορία ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ήτρε 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήτρε 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεβε 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε την τροπολογία 48. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ήτρε 8 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την Ήτρε 8. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε τη 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Γίνονται περίεργες συμμαχίες σε αυτή τη ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58, 59 και άγρι 7. Όχι, καταπίπτει. Άγρι 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62, καταπίπτει. 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήτρε 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την Ήτρε 13. Αρχή της ψηφοφορίας, πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 85. Πέρα τη ψηφοφορία. Όντω απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 86. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρα 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρα 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρα 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. δβ 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. δβ 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, να ελέγξουμε την δβ 9. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, Ο Υπουργό έρχεται στι 11, οπότε θα πρέπει να διακόψουμε. Λίγη η ηλεκτρονική ψηφοφορία και το επόμενο σημείο είναι η παρέμβαση του Εστονού Υπουργού Περιβάλλοντος. Φτάνει στις 11, άρα θα πρέπει να διακόψουμε μέχρι τότε.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 κολλάει. Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 Καλησπέρα σα. αγαπητοί συνάδελφοι. Or uh, ε, όχι καλησπέρα, δεν είναι ακριβώ απόγευμα, Τέλο πάντων. Παραδρομή. Καθίστε παρακαλώ. Το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Εστονική Προεδρία με τον κύριο Σιμ Κίσλερ, που είναι Υπουργό Περιβάλλοντος της Εστονίας. Ήρθε εδώ στα πλαίσια των ανταλλαγών απόψεων με τη νέα Προεδρία για να συζητήσουμε τις προτεραιότητες για το επόμενο εξάμεινο. Ψηφίσαμε για το ETS Υπουργέ σήμερα και την αεροπορία καθώς και για τη Λούλου CF. Με χαρά σας τον Αγγέλο. Ελπίζω κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας να δώσετε σημασία σε αυτά τα σημαντικά θέματα του περιβάλλοντος και τα θέματα της κλιματικής πολιτικής. Έχουμε διάφορα ζητήματα, διάφορους φακέλους που εκκρεμούν και ελπίζουμε να υπάρξει καλή συνεργασία μαζί σας, ούτως ώστε να προωθηθούν αυτά τα σημαντικά νομοθετήματα. Καλώς ήρθατε ακόμα μια φορά. Έχετε το λόγο για να μας μιλήσετε για τις προτεραιότητες προεδρίας σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ ικανοποιημένο που είμαι εδώ ενώπιον της Επιτροπής σας για να συζητήσουμε πώς θα μπορούσαμε μαζί να προωθήσουμε την περιβαλλοντική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίσουμε την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών, εξασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητε μας παραμένουν εντός των οικολογικών ορίων που επιβάλλει ο πλανήτης μας. Η Εστονία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε το προνόμιο να ασκούμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούμε ότι είναι μεγάλη μας τιμή και για να γιορτάσω την ιστορική αυτή περίσταση θα ήθελα να πω δύο λόγια στην μητρική μου γλώσσα, τα εστονικά. Στις αρχές της επόμενης χρονιάς η Εστονία θα γιορτάσει την εκατοστή επέτειο της ανεξαρτησίας της. Η μοίρα μας τα φύλαξε έτσι, ούτως ώστε να κάνουμε την Προεδρία έξι μήνες νωρίτερα από τα 100 χρόνια. Χαιρόμαστε για την πρόκληση αυτή που αναλαμβάνουμε. Ελπίζω να δράσουμε αποφασιστικότητα, ό,τι και αν συμβεί, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, για το κοινό μας στόχο και την ε, ευημερία μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε όλες τις σημαντικές προτάσεις ε, αποτελεσματικά και επικοδομητικά. Και τώρα θα συνεχίσω στα αγγλικά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πληθυσμού. Σήμερα υπάρχουν στον πλανήτη 7,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Με βάση τις πιο πρόσφατες ε, εκτιμήσεις του ΟΗΕ, θα φτάσουμε τα 10 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050. Και αυτό είναι μια καταστροφική προοπτική, αν συνεχίσουμε με τα σημερινά μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης. Ευτυχώς η Ευρώπη μεταβαίνει προς ε, μια κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και πιο αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, θα ήθελα να πω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θεωρούμε το Κοινοβούλιο ουσιαστικό εταίρο στην νομοθετική διαδικασία και προσβλέπουμε σε μια παραγωγική συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε επικοδομητικό διάλογο για να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατές ε, ρυθμιστικές και κανονιστικέ λύσει. Οι προτεραιότητε μα για το Συμβούλιο περιβάλλοντο καλύπτουν ε, τρία θέματα. Κλιματική αλλαγή, κυκλική οικονομία και οικολογική καινοτομία. Σημειώστε ότι θέματα που συνδέονται με τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων θα εξεταστούν σήμερα αργότερα από τον συνάδελφό μου Γευγένη Οσινόφσκι που είναι Υπουργό Υγεία και Εργασία στη χώρα μου. Οι προτάσεις ε, για τις οποίες θα σας μιλήσω έχουν συμπεριληφθεί ως θέματα προτεραιότητας στην Ευρωπαϊκή Νομοθετική Ατζέντα του 2017. Η Εστονία είναι έτοιμη να βασιστεί στην πρόοδο που σημείωσε η Μαλτέζικη Προεδρία και να προχωρήσουμε τον δόν περισσότερο σε όλα τα θέματα που είναι αυτή τη στιγμή επιτάπητος. Οι δράσεις για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή είναι το πιο πιεστικό θέμα στις προτεραιότητές μας. Η Εστονική Προεδρία εργάζεται εργοδός για να περάσει τις προτάσεις για το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 για το κλίμα και την ενέργεια που θα μας δώσει τη δυνατότητα να μειώσουμε τα, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% την επόμενη δεκαετία. Θα ξεκινήσω με τον ακροκονία ολίθο της κλιματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ETS, το Σύστημα Ανταλλαγής Εκπομπών. Τώρα που υπάρχει δυναμική θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με πιο παραγωγικό τρόπο οι προοπτικές είναι καλές, γιατί έχουμε τους ίδιους ε, στόχους, ένα ισχυρό ETS, το οποίο είναι κατάλληλο για αυτά που θέλουμε να κάνουμε και θα μας οδηγήσει στην υλοποίηση των στόχων του 2030. Σε ό,τι αφορά τις εκπομπές της αεροπορίας, σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε και ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε τους τριμερείς διαλόγους. Είναι κατάλληλη στιγμή τώρα να σας συγχαρώ για την ε, επιτυχή ψηφοφορία σήμερα το πρωί. Από πλευρά μα, η Μαλτέζικη Προεδρία πρέπει να σα πω ότι εξασφάλισε τη διαπραγματευτική εντολή τον Ιούνιο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τι συζητήσει με το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν. Το να επιτύχουμε μια συμφωνία είναι κρίσιμη σημασία για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για τι αεροπορικέ εταιρείε και να δείξουμε την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση προς, το, προς, τα, προς ένα παγκόσμιο μέτρο ε, που σχεδιάζεται υπό την συμφωνία για την διεθνή, της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας. Υπάρχει λοιπόν η δυναμική και περιμένουμε ε, και προσβλέπουμε σε μια επικοδομητική συνεργασία με την εισηγήτριά σας, την κυρία Τζούλι Γκέρλινγκ, και για τις δύο προτάσεις ETS. Επίσης, σας ευχαριστώ που επισκεφθήκατε την Εστονία το Μάιο και συναντήσατε την ομάδα μας, κυρία Γκέρλινγκ. Τώρα, αν δούμε τους τομείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ETS, και σε, αυτά, σε αυτούς τους τομείς υπάρχει σημαντική πρόοδος από το Κοινοβούλιο. Συγχαίρω τον εισηγητή, τον κύριο Γερμπράντη, που εξασφάλισε την εντολή για τους τριμερείς διαλόγους, για τον κανονισμό, για τον επιμερισμό της προσπάθειας. Επίσης, πάνω στο κανονισμό Λουσία έγινε θαυμάσια δουλειά υπό την αιγίδα του εισηγητή Νόρμπερτ Λίνς. Και συγχαρητήρια για την επιτυχή ψήφο σήμερα το πρωί. Από πλευράς μας, Προσπαθούμε να επιτύχουμε συμβασμό στο Συμβούλιο. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε τον Οκτώβριο στη γενική προσέγγιση και να ξεκινήσουμε τους του διαλόγους πριν τελειώσει η Προεδρία μας. Θα κλείσω την, τα θέματα της κλιματικής αλλαγής μιλώντας για τα θέματα των διεθνών διαπραγματεύσεων. Η Ευρώπη έπαιξε βασικό ρόλο για να επιτευχθεί η Συμφωνία του Παρισιού και έχουμε έκτοτε διατρανώσει τη δέσμευσή μας ο κόσμος έχει στραμμένο το βλέμμα προς την Ευρώπη για να, δείξει ηγετικό ρόλο, να παίξει ηγετικό ρόλο για την εφαρμογή της ατζέντα του Παρισιού. Το, το Νοέμβριο θα έχουμε την COP23 και θα είναι σημαντικό, σημαντική εκδήλωση καθώς η δράση για την κλιματική αλλαγή έχει μπει σε, αποφασιστικό, σε αποφασιστική τροχιά. Η Προεδρία μας είναι εστιασμένη στην υλοποίηση του προγράμματος ε, του Παρισιού και στο να τεθούν οι προϋποθέσεις για να διευκολυνθεί ο διάλογος το 18. Θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα σε μια τύπη υπουργική συνάντηση στο Τάλιν. Το βασικό δεύτερο σημείο του προγράμματος της Προεδρίας είναι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης του πακέτου για τα απόβλητα που θα είναι η βάση για να υπάρξει μια ε, κυκλική οικονομία που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους φυσικούς πόρους. Η Προεδρία μας αναγνωρίζει την τεχνική φύση του πακέτου και προσπαθούμε να επιτύχουμε μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγητή, την κυρία Σιμώνα Μποναφέ, για την εντυπωσιακή δουλειά που έκανε σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο πακέτο προτάσεων παράλληλα. Προσβλέπουμε επίσης στις επερχόμενες προτάσεις της Κομισιόν που θα είναι ουσιαστικά η επόμενη φάση, το επόμενο βήμα στο πακέτο της κυκλικής οικονομίας, προτάσεις για τα πλαστικά, την επαναχρησιμοποίηση των λιμάτων και την διαπαφή για τα χημικά προϊόντα, ε, την ομοθεσία για τα προϊόντα και απόβλητα που περιμένουμε αργότερα το 2017. Επίσης, τονίζουμε το ρόλο της οικολογικής καινοτομίας για να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια κυκλική οικονομία. Είναι κοινή προτεραιότητα για το τρίο των Προεδριών, στο οποίο συμμετέχει η Βουλγαρία και η Αυστρία. Μαζί θέλουμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε, να βοηθήσουμε, τόσο να προωθήσουμε το θέμα αυτό στην, ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Πέμπτη θα κάνουμε μια άτυπη υπουργική συνάντηση στο, στο Ταλίν, όπου θα επικεντρωθούμε στην διαφάνεια για τα προϊόντα, στι έξυπνε πόλει και στην χρηματοδότηση τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το μήνα του Οκτωβρίου θα τον αφιερώσουμε στην οικολογική καινοτομία και θα διοργανώσουμε διάφορε εκδηλώσει που θα διερευνούν ψηφιακέ ε, λύσει και λύσει που θα βασίζονται στη φύση. Τελικά θέλουμε να υιοθετήσουμε το Δεκέμβριο τα συμπεράσματα του Συμβουλίου το 2018 τελειώσει και το τρίο των δικών μας προεδριών και ελπίζουμε μέχρι τότε να έχουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για μία συνεκτική πολιτική για τα προϊόντα. Επίσης, θέλουμε να ενισχύσουμε το ρόλο των καταναλωτών και να συμπεριλάβουμε εδώ και το δημόσιο τομέα που θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη ζήτηση, να ζητήσει να υπάρχουν περισσότερες οικολογικές ε, καινοτόμες λύσεις μέσω ε, προμηθειών πράσινων και κυκλικών. Η εστίασή μας στην οικολογική καινοτομία ευθυγραμμίζεται με τους ευρύτερους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης όπως τονίζονται στην ατζέντα του 2030. Καλωσορίζουμε τη θετική και δραστήρια στάση του Κοινοβουλίου και το πρόσφατο ψήφισμα για το θέμα αυτό. Εκτιμούμε την πρωτοβουλία που έδειξε ο εισηγητής Σεμπ για το θέμα αυτό. Το Συμβούλιο υιοθέτησε τα συμπεράσματά του τον Ιούνιο και περιμένουμε να υπάρξει περαιτέρω δράση από πλευρά Κομισιόν πια για να εντοπίσουμε τα κενά στην ευρωπαϊκή πολιτική και να προτείνουμε μια στρατηγική για την εφαρμογή της. Κλείνοντας την ε, παρουσίασή μου, θα ήθελα να σας πω ότι πάνω απ' όλα η Εστονική Προεδρία ελπίζει να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος πάνω στις προτάσεις για το σύστημα ETS της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει το σύστημα μείωσης των εκπομπών και το πακέτο για τα απόβλητα. Επίσης, θεωρούμε τα μέλη αυτής της Επιτροπής πολύτιμους εταίρους για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, κυρίες και κύριοι. Περιμένω τα σχόλιά σας. Thank Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, για την εισήγησή σας. Πριν να αρχίσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να πω ότι ότι ο κύριος Νένο που είναι Υπουργός Βιομηχανίας της Βουλγαρίας, είναι σήμερα μαζί μας και μάλλον προετοιμάζεται για την επόμενη Προεδρία του Συμβουλίου που την αναλαμβάνει η Βουλγαρία. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και εσάς και αρχίζουμε με ερωτήσεις, καταρχήν από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Λίζα έχει το λόγο από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, για τη δουλειά που καταβάλλετε και για την παρέμβαση που κάνετε σήμερα εδώ. Ε, υποστηρίζουμε αυτέ τι απόψεις ε, και αυτό που μας είπατε, ότι θέτε την προστασία του κλίματος σε προτεραιότητα της προεδρία σα. Ε, θέλουμε φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα, ιδίως μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ. Αυτή είναι σαφώ και η θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, αλλά παράλληλα θέλουμε η βιομηχανία που ασχολείται με την τελευταία λέξη τη τεχνολογία να μην εκδιωχθεί από την Ευρώπη. Και γι' αυτό θέλουμε να βρούμε μια σωστή λύση στον τριμερή διάλογο ε, για το ETS. το Κοινοβούλιο θέλει κατευθείαν στην αρχή της επομένης περίοδου να ξεκινήσουμε με τα πιστοποιητικά. Συζητήθηκε ένας αριθμός 300 εκατομμυρίων ε, πιστοποιητικών ε, και για το θέμα της ε, προστασίας είναι πολύ σημαντικό να μην μας διαφύγει η δυνατότητα μιας ποιοτική αξιολόγησης. Και θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των πιστοποιητικών που δεν έχουν κόστος. Παραμένει σημαντικό το ποσοστό για τη δική μου πολιτική ομάδα και να μην παραμείνει το Συμβούλιο στο 2% να φτάσουμε στο 5%. Έχουμε την έκθεση της κυρίας ε, Γκέρλινγκ, την οποία μόλις εγκρίναμε, για τις ε, αεροπορικές, ε, για τις εκπομπές στις αεροπορικές μεταφορές και θα πρέπει να συνδέσουμε διάφορους τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεγαλύτερες φιλοδοξίες στον ένα τομέα μπορούν να συνδυαστούν και με τους άλλους τομείς. Η επιστημονική υπηρεσία του Κοινοβουλίου Μίλησε για το 1% των πιστοποιητικών. Ε, το 1% είναι μεγάλο ποσοστό όταν ξέρουμε ότι η διαφωνία είναι από το 2% στο 5%. Και για το LULUCF και για τον επιμερισμό προσπαθειών, ως ε, Προεδρεύων του Συμβουλίου θα πρέπει να φροντίσετε να μην αποδυναμωθεί η θέση μας και για το Παρίσι και για τις διεθνείς ε, συζητήσεις. Μερικές φορές γίνεται επικίνδυνη αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Um, η κυρία Νταλή από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ε, χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε ότι η Εστονική Προεδρία είναι πολύ φιλόδοξη για το ε, μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπει και καινοτόμα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Διέτρεξα το πρόγραμμά σας Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, εμείς οι σοσιαλιστές και δημοκράτες συμφωνούμε ότι θα πρέπει να μειώσουμε τα αέρια θερμοκηπίου όπως συμφωνήθηκε από τη Συμφωνία των Παρισίων και θα πρέπει τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οδηγήσουν σε ένα προοδευτικό και φιλόδοξο σχέδιο και να μην έχουμε μόνο ωραία λόγια στο χαρτί. Τώρα με βάση το ίδιο σας το πρόγραμμα και με, την, και βάση την εισήγησή σας είναι πολύ θετικό ότι είπατε ότι στην αεροπλοεία, στο πρόγραμμα ETS, θέλετε να φτάσουμε σε αυτά συμπεράσματα για το ETS στην αεροπλοεία και να ολοκληρωθεί το θέμα υπό την Προεδρία σας. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει σπουδή στο θέμα. Μιλήσατε και για την αγορά των οδικών μεταφορών. Θα εργαστείτε και επ' αυτής. Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος από εσάς και στο πρόγραμμά σας Μιλήσατε για αρχή συζητήσαν για να προβάλλουμε ε, οικολογικές και καινοτόμες ε, λύσεις για την ε, κυκλική οικονομία. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας μιλήσετε για λεπτομέρειες για να έχουμε καλύτερα στοιχεία για το ποιες είναι οι προτάσεις σας επί του θέματος. Ευχαριστώ. Η κυρία τώρα από το ECR. Ευχαριστώ, θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον ε, Υπουργό στην Επιτροπή μας σήμερα. Οι προτάσεις που με ενδιαφέρουν αφορούν τις ανταλλαγές εκπομπών αερίων, το ETS. Και η Εστονική Προεδρία ε, έχει αναλυφθεί εδώ και μία εβδομάδα και παρόλα αυτά έχουμε ασχοληθεί με αρκετά θέματα. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σπουδή που δείχνουμε επί του θέματος, αν και δεν έχουμε προβεί σε ολοκληρωμένη αντιστροφή πορείας, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, αεροπλοεία και το ETS θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα του ETS της αεροπλοείας και θα ήθελα να προχωρήσουμε παράλληλα έτσι ώστε, να τελειώσουν και τα δύο την ίδια χρονική στιγμή. Ο Πίτερ Λίζε αναφέρθηκε σε αυτά τα στοιχεία σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα που διέπει τα δύο συστήματα και δεν χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Έχουμε τις διαφορές μας και δεν έχει νόημα να παρατείνουμε και να κολλησιεργούμε. Σέβομαι το γεγονός ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές ως προς την εντολή μας και αυτό δεν μπορεί να γίνει εν μία νυχτή. Υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν επιπτώσεις ε, και στην οικονομία και στο περιβάλλον. Σας, και, σας εύχομαι κάθε ε, επιτυχία και ελπίζω να συνδράμουμε σε αυτό. Ε, έχω ένα ερώτημα να υποβάλω, γιατί τα άλλα τα καλύψατε. Μιλήσατε για συνέργεια των πακέτων, γιατί είπαμε ότι δεν έχουμε τα δύο ETS μόνο, αλλά και το Λουλουσιεφ, τον επιμερισμό προσπαθειών και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι τα λιγό, το λιγότερο επιτυχές στοιχείο είναι ο συντονισμός και η συνέργεια αυτών των πακέτων για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε στο σύνολό τους γιατί υπάρχει ρήξη από τον ένα ή τον άλλο τομέα. Αυτή είναι μια ευκαιρία για σας και δεν ξέρω πώς μπορούμε να φτάσουμε σε ένα συνολικό πακέτο μέχρι το τέλος της όλης διαδικασίας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκέρλ, ο κύριος Χερμπράντι από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον ε, Υπουργό Κίσλερ που ήρθε εδώ να μας παρουσιάσει το εξαμηνιαίο πρόγραμμά του. Προσβλέπω στην επιτυχία του, της Προεδρίας σας, γιατί είδα και την ιστοσελίδα σας και έλαβα και αυτή, αυτά το, τη σακούλα, η οποία έχει στοιχεία, πράσινα στοιχεία, αλλά άμα την αναποδογυρίσετε είναι εντελώς πράσινη. Ελπίζω λοιπόν ότι το πρόγραμμά σας φαίνε, φαίνεται να έχει πράσινα στοιχεία εδώ και από εκεί, αλλά αν το ε, αναποδογυρίσουμε βλέπουμε ότι είναι απόλυτα πράσινο ως προς την ε, βιοπικιλότητα. Ξέρουμε ότι δεν θα φτάσουμε στο, στους στόχους του 2020 ως προς την ε, στρατηγική βιοπικιλότητας η Επιτροπή έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά τα κράτη-μέλη σιωπούν. Τι θα κάνετε λοιπόν κατά την Προεδρία σας για να χρησιμοποιήσετε αυτό το έμβλημα που έχετε, την καρδερίνα, για να πείσετε τους συναδέλφους να επιταχύνουν ε, του στόχους μέχρι το 2020 όσον αφορά την βιοπικιλότητα και τη γεωργία. Τώρα, ως προς το κλίμα, και στον επιμερισμό προσπαθειών και ευθυνών. Ξέρουμε τι συμβαίνει στον κόσμο με τον Τραμπ, την Τουρκία και την αλλαγή της άποψής του ως προς το Παρίσι. Άρα θα πρέπει να παραμείνουμε στην πορεία μας και όταν ε, συμβεί η επόμενη έκρηξη να έχουμε το δικό μας μήνυμα. Δηλαδή, εάν στον οκτώ, τον Οκτώβριο στο ε, Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος φτάσουμε σε έναν απτό στόχο, θα πρέπει να δούμε πώς θα τον προωθήσουμε. Άρα η ερώτησή μου είναι, επειδή Οκτώβριος δεν είναι και πολύ μακριά, τι θα κάνετε ως προς τα κλιματικά και τον επιμερισμό προσπαθειών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κονέτσνα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώ ήρθατε στη σημερινή μα συνάντηση. Χαίρομαι ιδιαίτερω που είχατε την ε, δυνατότητα να μα επισκεφτείτε. Και χαίρομαι που έχουμε και εκπρόσωπο τη επόμενη στη σειρά Προεδρία τη Βουλγαρία. Θα ήθελα όλες οι προτεραιότητες να ευοδοθούν αυτές που αναφέρετε, αλλά η πολιτική είναι η τέχνη του να επιτυγχάνουμε το εφικτό και όλοι συμφωνούμε από αυτού. Υπάρχουν τόσα πολλά θέματα προς συζήτηση, τα οποία είναι και αλληλοσυνδεόμενα. που νομίζω ότι θα ολοκληρωθούν υπό την επόμενη Προεδρία και θα συνεχίσουμε ε, με τα ίδια θέματα. Άρα η ε, συνέχεια είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, συνέχεια. Όπως και οι συνάδελφες, και εγώ πιστεύω και αυτό έδειξε και ο τριμερής διάλογος χθε, ότι ίσως μπορούμε να ολοκληρώσουμε τον τριμερή διάλογο για το ETS και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί για διάφορους λόγους έχει καθυστερήσει για κάποιο διάστημα και για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το ETS και να έχουμε μια συνολική προσέγγιση για το LULUCF και τον, και τον επιμερισμό προσπαθειών θα είναι σημαντικό να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και στη δική σας Προεδρία. Η ερώτησή μου είναι Πώς βλέπετε τα ενεργειακά θέματα, διότι εδώ έχουμε περισσότερο έντονες ε, αντιπαραθέσεις. Ε, όλοι Καταλαβαίνουμε τις προτεραιότητές σας λόγω και της γεωπολιτικής σας θέσης και κατά την παρουσίασή σας είπατε ότι θέλετε να ε, καταλήξουμε σε ένα βελτιωμένο τρόπο διασύνδεσης ε, του δικτύου στην Ευρώπη και ότι πρέπει να συνεισφέρουμε στη σύνδεση βορρά-νότου. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς προτίθεστε να προχωρήσετε και αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ο κ. Σάικχαουτ. Ευχαριστώ τον Υπουργό που μα μίλησε για αυτό το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Δεν έχω δει ποτέ τόσους πολλούς ε, νομοθετικούς ε, φακέλους ε, στα πλαίσια μιας προεδρίας. Έχουμε, σε μια σύντομη προεδρία, γιατί έχουμε τέσσερις μήνες. Έχουμε το κλιματικό πακέτο, το ενεργειακό πακέτο, που δεν νομίζω ότι αφορά μόνο τους Υπουργούς Ενέργειας και ελπίζω να παίξετε και εσείς το ρόλο σας και για αυτό το θέμα, γιατί όπως είπε ο κυρία Κονέτσκα, ε, δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε τα θέματα ενέργειας μόνο στους υπουργούς ενέργειας. Ε, και υπάρχει στη Βόνη η επόμενη σύνοδος κορυφής για το κλίμα. Ε, και υπάρχει και το ETS. Σας ευχαριστώ για την πολύ ισχυρή δέσμευση για την Συμφωνία του Παρισιού μετά την αποχώρηση του Τραμπ. Ε, χαίρομαι γι' αυτό, αλλά έχω ένα θέμα, ένα πρόβλημα αξιοπιστίας εδώ. Γιατί αν η Ευρώπη κάθε φορά ε, μιλάει για την σημασία της εφαρμογής του Παρισιού, ε, τότε θα μας κάνουν την ερώτηση για να απαντήσουμε στο εξή ερώτημα. Ε, τι κάνει η Ευρώπη για να εφαρμόσει την ε, συμφωνία του, του Παρισιού στην Ευρώπη. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Λούλου Σιέφ, ας πούμε. Ελπίζω τον Οκτώβριο το Συμβούλιο να συμφωνήσει και, να συμφωνήσει και για τον επιμερισμό προσπάθειας. Αλλά ξέρουμε ότι σε μια διαπραγμάτευση υπάρχουν διάφορα κόλπα που παίζονται ε, με, το πώς υπολογίζουμε, πώς υπολογίζουμε. Ε, μην ξεχνάτε ότι έχει ένα, μία δεξαμηνή ε, απομείωση η Ευρώπη. Ε, το άρθρο 5 ε, της Συμφωνίας του Παρισιού, να σας το διαβάσω, βοηθάει, λέει. Τα μέρη θα πρέπει να λάβουν δράση για να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις ε, δεξαμενές και τα αποθετήρια ε, αερίων του θερμοκηπίου. Πώς θα συμμορφωθεί η Ευρώπη με το άρθρο αυτό εάν δεν έχουμε σωστό σύστημα καταμέτρησης ας πούμε. Σας παρακαλώ η συμφωνία Λουλουσιέφ εξασφαλίστε το να μην έχει παραθυράκια. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να σεβαστούμε το άρθρο 5 της συμφωνίας του Παρισιού. Γιατί όχι, πιστεύω ότι θα έχουμε πρόβλημα αξιοπιστίας γιατί θα κατηγορούμε τον Τραμπ, αλλά εμεί δεν θα εφαρμόζουμε στο εσωτερικό μα το, τη Συμφωνία του Παρισιού. Ευχαριστώ τον, τον κύριο Έικχαουτ. Η κυρία Ντορνάνο από το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την παρουσία σας. Επιλέξατε να επικεντρώσετε τις δράσεις σας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ε, αλλά μιλάτε αποκλειστικά και τη Συμφωνία του Παρισιού. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ και μήνες εστιάζουμε τις συζητήσεις μας σε αυτή τη συμφωνία και καταδικάζοντας την περιβαλλοντική πολιτική του Ντόναλτ Τραμπ. Όμως είναι και η ώρα να λάβουμε υπόψη την ε, αποχώρηση του, των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού και να δούμε τι συνέπειες έχει. Επίσης, να σας ρωτήσω, θα προωθήσετε μια νέα διεθνή δράση στα πλαίσια των συμφωνιών ε, και των οργανισμών που είναι μέλη και είπα, παραδείγματο χάρη, η σύμβαση πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, κλιματική αλλαγή OMI, ε, OSAE, ε, που νομιμοποιούνται η κάθε μία με βάση αρμοδιότητες της να δρά κατά της κλιματικής αλλαγής. Μία από τις βασικές ε, προτεραιότητες της Προεδρίας σας είναι να προωθήσει επίσης την κυκλική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, θέλετε πραγματική βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων. Ελπίζω η Εστονία θα προτείνει θέμα, ε, συγκεκριμένα πράγματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι και η δική σας πρωτεύουσα το Τάλιν ε, διακρίθηκε μέσα από μια φιλόδοξη πολιτική τα τελευταία χρόνια. Ποιες είναι οι καλές πρακτικές που θα μοιραστείτε με τα άλλα κράτη-μέλη ό,τι αφορά την επεξεργασία των αποβλήτων. Ευχαριστώ. Μάλιστα, κλείνουμε έτσι τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ο Υπουργό θα απαντήσει. Thank you, ladies and gentlemen. Um, I we will take into account all your, all your uh, remarks. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σημείωσα όλες σας τις παρατηρήσεις. Βλέπετε ότι είναι φιλόδοξο το πρόγραμμά μας και αναγνωρίζουμε όλα τα πολύπλοκα νομικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Σας διαβεβαιώνω ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια στο Συμβούλιο των Υπουργών και νομίζω ένα γενικότερο ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε διμερείς συναντήσεις, να κάνουμε συζητήσεις με όλα τα κράτη-μέλη, για να βρούμε τη σωστή λύση. Αυτό ισχύει και για τη διαδικασία του τριμερούς διαλόγου. Πρέπει να βρούμε το χρόνο και να καταβάλουμε τις απαραίτητες προσπάθειες. Περνώ τώρα στις συγκεκριμένες σας ερωτήσεις. Ο κύριος Λίζα καταρχήν, που μίλησε για την κλιματική αλλαγή με το ETS και την αεροπορία. Όπως είπα ήδη, έχουμε διασφαλίσει την εντολή διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι τον Ιούνιο υπό Προεδρίας της Μάλτας. Και νομίζω ότι θα έχουμε σύντομη πρόοδο στο θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντική η συμφωνία για όλους ε, τους ε, εμπλεκομένους και για να δείξουμε ότι όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται για να έχουμε πριν από το 2021 μετρήσεις με βάση ε, την αγορά και στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Θέλουμε να διατηρήσουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, αναγνωρίζοντας παράλληλα τους κινδύνους που υφίστανται για κάποιους κλάδους, γιατί και η βιομηχανία θέλει να συμβαδίζει με τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Η κυρία Νταλή και η κυρία Γκέρλινγκ έκαναν επίσης ερωτήσεις για τα θέματα του κλίματος. Όπως ήδη σας είπα, θέλουμε να έχουμε μία ισορροπημένη διαδικασία για το ETS και για το LULUCF. Θέλουμε να προχωρήσουμε και στους δύο τομείς. Και μαζί με την πρόταση για την αναθεώρηση του συστήματος ETS, Είναι ζωτική σημασία οι προτάσεις εν ώψη του συνολικού πλαισίου για την ενέργεια. Έχετε δίκιο κυρία Γκέρλινγκ, υπάρχει συνέργεια μεταξύ των ενεργειακών θεμάτων και στις διαπραγματεύσεις μας αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι σύνθετες οι λύσεις που πρέπει να βρεθούν. Προς τον κύριο Άικαουτ. Εσείς κάνατε πιο συγκεκριμένα ερωτήσεις για το Λουλουσιεφ. Η Προεδρία μας, όπως σας ανέφερα, θα ασχοληθεί εντατικά με το σχέδιο κανονισμού Λουλουσιεφ και μαζί με τον κανονισμό για το ETS και τον επιμερισμό προσπαθειών Μπορούμε να προχωρήσουμε και στην πρόταση για το Λουλουσιεύ και να προωθήσουμε τις δεσμεύσεις μας, τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού. Κατά τις διαπραγματεύσεις προσπαθούμε και να βρούμε ισορροπημένη λύση και να παραμείνουμε φιλόδοξοι. Είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε συγκεκριμένα ε, τεχνικά στοιχεία και υπολογιστικά στοιχεία και οι υπολογισμοί μας θα πρέπει να υποστηρίζουν το στόχο μας. Θα κάνουμε λοιπόν κάθε προσπάθεια να εκπληρώσουμε σωστά το ρόλο μας. Mr. and Mr. Eichhout uh, pointed out the... Ο κύριος Γκέρμπραντι και ο κύριος Eichhout τόνισαν τη σημασία των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ αποτελούν ε, ένα μεγάλο πλήγμα στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Μα ενθαρρύνει όμως η απάντηση της διεθνούς κοινότητας συμπεριλαμβανομένη τη ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών τη, αλλά και των επιχειρήσεων και άλλων εμπλεκομένων, οι οποίοι όλοι δήλωσαν εκ νέου την ισχυρά δέσμευσή τους για τη διαδικασία του Παρισιού και μεμονωμένες πολιτείες ή και πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν δηλώσει την υποστήριξή τους για μείωση εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακος. Όσον αφορά την COP23 στη Βόνη, θα φροντίσουμε να διασφαλίσουμε τη σημαντική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσουμε την Συμφωνία του Παρισιού και όλα τα σχετικά στοιχεία. Και μια επιτυχημένη συνεδρία του Συμβουλίου τον Οκτώβριο θα είναι κλειδί για αυτή τη διαδικασία. Κυρία Ντονανό. έκανε μια ερώτηση για τη δέσμη μέτρων για τα απόβλητα. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο, ούτως ώστε μέχρι το τέλος του έτους να καταλήξουμε σε μια πολιτική συμφωνία. Υπάρχουν καλές πρακτικές για την διαχείριση των αποβλήτων. τις οποίες ε, έχουμε υιοθετήσει στην Εσθονία και μπορούμε να τις μοιραστούμε και με άλλες χώρες. Ήδη από το 2005 έχουμε ένα σύστημα το οποίο το εφαρμόζουμε για την απόθεση αποβλήτων και έχουν επισκεφθεί την Εστονία πολλά κρατημέλη και πολλοί ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούσαν να διδαχθούν από το δικό μας σύστημα και τον τρόπο με τον οποίο το έχουμε οργανώσει. Ο κύριος και η κυρία Κανίτσινα ρώτησαν για την χειμερινή δέσμη μέτρων ε, για τα ενεργειακά θέματα. Η Εστονική Προεδρία ε, θα διασφαλίσει μια ισορροπημένη και αποτελεσματική νομοθεσία και ο σκοπός μας είναι να επιτύχουμε πρακτικά αποτελέσματα επαυξάνοντας το έργο που έχει ήδη η Προεδρία της Μάλτας. Θα προχωρήσουμε με τη δέσμη μέτρων για την ε, καθαρή ενέργεια τονίζοντας το σχεδιασμό της αγοράς ε, ηλεκτρισμού που αποτελεί βασικό σημείο της Ενεργειακής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα προχωράμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Η κυρία Σερ Πέρεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία και το Συμβούλιο γιατί ήρθαν σήμερα. Έχω μία ερώτηση που έχει επίγοντα χαρακτήρα. Στις 6 ε, Ιουνίου 17 είχαμε ένα πρόγραμμα δράσης για τις ε, προτεραιότητες για την εφαρμογή του Nature και των ε, οικολογικών προδιαγραφών. Έχουμε και το σχέδιο βιωσιμότητας στη Βόρειο Θάλασσα. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την ε, πρόκληση η Προεδρία σε σχέση με τους περιορισμούς στη Γεωργία και την αλληλεία και ιδιαίτερα σε σχέση με την ε, αλίευση τόνου που είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό σχέδιο και Υπάρχει μελέτη βιωσιμότητας από ό,τι άκουσα μέσα στα πλαίσια του Nature κάτι τέτοιο είναι εφικτό, αλλά έχετε μία επαφή με τους ε, αλληλείς ε, επί του θέματος. Εμείς θα μεταβούμε στη Γερμανία με την Επιτροπή Αλληλείας για να αποτιμήσουμε το όλο θέμα και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θέλουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε υπέρ της ε, φύσης ε, και της οικολογίας, αλλά δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, γιατί υπάρχει μία οικονομική και κοινωνική διάσταση και πολλές φορές αυτή την ε, Επιτροπή δεν λαμβάνουμε τόσο υπόψη αυτές τις πτυχές. Ο κύριος Πάρνιο έχει το λόγο, αντιπρόεδρος. Κύριε Υπουργέ, όπως είπατε και στην εισήγησή σας, οι έξι αυτοί οι μήνες της Προεδρίας θα είναι πολύ σημαντικοί για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, όχι μόνο για την COP23 στη Βόνη τον Νοέμβριο, αλλά και τη διάσκεψη των Παρισίων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν κατά τη τελευταία διάσκεψη των G20. Σε αυτή την κρίσιμη λοιπόν περίοδο, όπως υπενθυμίσατε, ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να αποσυρθεί από τη Συμφωνία των Παρισίων παρά την ομόφωνη αντίδραση του κόσμου για την απόφαση αυτή. Ξέρουμε ότι ακολουθεί μια πολιτική προστατευτισμού και απομονωτισμού και αυτό αφορά 30 ε, πολιτείες των ε, Αμερικανών που αντιτάσσονται στην απόφαση του Ντόναλτ Τραμπ. Η Εσθονική Προεδρία λοιπόν θα πρέπει να αναλάβει μία πρωτοβουλία έτσι ώστε υπό το φως του COP, ε, της COP23 και της διάσκεψης των Παρισίων να ε, λάβει κοινέ αποφάσεις με τις Αμερικανικές πολιτείες, τις επιχειρήσεις και τις πόλεις που αποφάσισαν να παραμείνουν στη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Μπάρακ Ομπάμα τον Δεκέμβριο του 2015. είναι τα σχέδιά σας έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος με τους Αμερικανούς που είναι υπέρμαχοι αυτή τη συμφωνία των Παρισίων μέσα στο επόμενο εξάμεινο. Σας ευχαριστώ. Πολύ η κυρία Γκέρλινγκ έχει το λόγο. Όχι, α, συγγνώμη. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. έχω μία ερώτηση ε, για ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε ε, για το τη διακυβέρνηση των ωκεανών που αποτελεί αντικείμενο μιας ε, ανακοίνωσης της Επιτροπής. Είναι σαν μια θάλασσα με μεγάλο μήκος ακτών ο ωκεανός. Ποια θα είναι η συνέχεια που θα δοθεί στην διάσκεψη για τους ωκεανούς Ε, τι προτεραιότητα δίνει η Προεδρία σας ε, στην ε, θάλασσα και στους ωκεανούς. Μας ενδιαφέρει όλους, ενδιαφέρει και τη χώρα σας, ενδιαφέρει τη Βαλτική. Μας ενδιαφέρουν ε, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος ε, και ε, μπορεί να έχει παρατηρηθεί μια βελτίωση σε σχέση με άλλες θάλασσες, γύρω στο 2%, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Ευχαριστώ πολύ. κύριος Εκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στην συνεδρίασή μας να μας μιλήσετε για το φιλόδοξο πρόγραμμά σας. Έχω μία ερώτηση. Με την έκθεση του συναδέλφου Σεπ Dance, ζητείτε από την Επιτροπή αλλά και από άλλους εμπλεκομένους να ασχοληθούν και με τις εκπομπές μεθανίου. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα, το μεθάνιο είναι 25 φορές πιο επιβλαβές από το διοξίδιο του άνθρακος και όλοι γνωρίζουμε ότι από ε, τις εκτεταμένες ε, ε, επιχειρήσεις εκτροφής ζώων προέρχονται μεγάλες εκπομπές μεθανίου. Έχετε πρόθεση να καταβάλλετε προσπάθειες για τη μείωση εκπομπών μεθανίου και θα είχατε το θάρρος όταν μιλάμε για μια τέτοια μείωση να συμπεριλάβετε και μια μείωση του ζωικού κεφαλαίου αυτό θα είχε ε, μεγαλύτερη ε, αποτελεσματικότητα και όσον αφορά την επιβάρυνση των υπογείων ε, υδάτων και για την βιοπικιλότητα. Η εντατική εκτροφή ζώων ξέρετε ότι είναι επιβλαβής για αυτούς τους τομείς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Φαρία. Uh, ευχαριστώ, κύριε Κίσλερ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σα ε, και σας ευχαριστώ για τη φιλοδεξία που δίνει η Προεδρία σας ε, προωθώντα την ατζέντα για το θέμα της κλιματική αλλαγή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, είπαν ότι σκοπεύουν να αποχωρήσουν από τη Συμφωνία του Παρισιού. Παρά τα όσα είπε ο συνάδελφος, Ε, ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές πολιτείες, παρά την άποψη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, έχουν διαφορετική άποψη. Το Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει τη στρατηγική για τα πλαστικά για να μειώσει τα πλαστικά στη θάλασσα. Ελπίζουμε ε, να έχουμε και το χρονοδιάγραμμα ε, για ένα ψήφισμα και συγκεκριμένα μέτρα καθώς και πολιτικές και εργαλεία. Το πρόβλημα είναι τόσο σημαντικό ε, που θέλει παγκόσμια απάντηση. Ε, κάθε λεπτό ε, πετιώνται στον ωκεανό και στη θάλασσα πάνω από ένα εκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια. Χρειάζεται απάντηση. Ω Υπουργό ε, Περιβάλλοντο μια παράκτεια χώρα, θα μπορούσατε να μα πείτε τα πολύ συγκεκριμένα μέτρα και προτεραιότητα τη Εσθονική Προεδρία, ούτω ώστε να συνεισφέρετε στην προστασία των ωκεανών μα και του θαλάσσιου περιβάλλοντο. Και τι θα πείτε στην Μάλτα τον επόμενο Οκτώβριο, στη διάσκεψη που θα γίνει για τους ωκεανούς. Ευχαριστώ κύριε Φαρία. κυρία Γκούταλαντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Πρωθυπουργέ που ήρθατε εδώ. Θέλω να πω δύο λόγια για το ETS, το σύστημα ανταλλαγής εκπομπών και την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κλιματική πολιτική σημαίνει ότι όλη η κοινωνία πρέπει να συνεισφέρει στην κοινή μας προσπάθεια για να καταπολεμήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Όλοι οι τομείς έχουν ευθύνη εδώ. Αυτό συμπεριλαμβάνει και το θαλάσσιο τομέα, που σήμερα είναι ο μοναδικός τομέας ο οποίος δεν έχει κανένα στόχο για τη μείωση της συνεισφοράς του στις εκπομπές. Όλες αυτές οι εκπομπές θα αυξηθούν κατά 250% με 200 μέχρι το 2050 από την ναυτιλία. Δεν είναι αποδεκτό αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο πρότεινε ότι και ο θαλάσσιο τομέα και η ναυτιλία θα πρέπει να ενταχθεί στο ETS. Εάν ο IMO δεν ετοιμάσει ένα επαρκές σύστημα μέχρι το 2023, ε, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Αυτό σημαίνει αλληλεγγύη. Κανένα δεν πρέπει να μείνει πίσω. Ε, το να περάσουμε σε μια βιώσιμη κοινωνία δεν μπορεί να αφήσει εκτός ε, περιοχές, εργαζόμενοι που πλήγησαν πιο πολύ από τη μετάβαση. Γι' αυτό το Κοινοβούλιο πρότεινε μια δίκαιη μετάβαση ε, υπέρ της ε, κινητικότητας της απασχόλησης, νέες επιχειρήσεις, ούτως ώστε κανένας να μην μείνει ξεχασμένος σε αυτή τη μετάβαση προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Το ερώτημά μου είναι πώς προωθεί το Συμβούλιο αυτά τα δύο πολύ σημαντικά θέματα στο πακέτο του ETS. Ο κύριος Λάινεν. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Γκερμπράντι έχει ήδη επενέσει το έργο σας. Εγώ επενώ και τη γραβάτα της Προεδρίας. Κάθε φορά μας δίνετε μια Προεδρία, η δική σας, γραβάτα όχι μόνο είναι χρήσιμη, αλλά και πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε για τα δώρα σας η COP23 θα είναι για σας ε, μια γενική δοκιμή, να δούμε και πώς αντιδρά, ε, αντιδρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ίσως και η Τουρκία. Θα χρειαστεί να σχηματίσετε και νέες συμμαχίες. Ε, πρέπει να διαμορφώσουμε μια συμμαχία των φιλοδόξων. Με ενδιαφέρον παρακολουθώ αυτά τα οποία προτείνεται για την οικοκαινοτομία η Εστονία θα μπορούσε να συνεισφέρει πολλά σε αυτόν τον τομέα. Και με το eco-design, με την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, έχουμε αναδείξει ε, τη σημασία του σωστού σχεδιασμού και υπάρχει μεγάλο δυναμικό σε αυτόν τον τομέα. Η ψηφιοποίηση των προϊόντων ε, και των υπηρεσιών θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στην Ευρώπη. Για την προστασία της φύσης θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει ένα σχέδιο δράσης, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα. Και η Προεδρία σας θα αρχίσει τη συζήτηση για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάτι θα πρέπει να φροντίσετε να πάρουν και η βιοπικιλότητα και η προστασία της φύσης. Θα πρέπει από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα να περάσουν κονδύλια, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη για αυτά τα σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βγάνεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας και ως ε, Βρετανός και Σοσιαλιστής χαίρομαι διπλά γιατί αν δεν ήμουν εγώ θα έπρεπε να ακούσετε, εδώ θα έπρεπε να ακούσω τον Μάικλ Γκόβ. Ψηφίσαμε για το LULUCF και υπήρχαν πολλοί που ήθελαν να κάνουν λιγότερο φιλόδοξη την πρόταση της Επιτροπής, αλλά εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος σαφώς ε, κερδίσαμε αυτή τη νίκη και για να ε, επιμείνω σε αυτά τα οποία ε, σε αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος από τους Πρασίνους, θέλω να σας παρακαλέσω να μην αποδυναμωθεί αυτή η πρόταση για το Λούλου Κάτι το οποίο προσπαθούμε να επιτύχουμε με υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων είναι να δοθούν κίνητρα για την ε, κατασκευή κτηρίων ε, από ξύλο ε, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσω του κανονισμού Λουλουσιεφ γιατί τα ξύλινα κτίρια δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακος όπως και τα δένδρα και υποκαθιστούν το χάλιβα και, ξέρουμε, και το τσιμέντο. Ξέρουμε ποιε είναι οι εκπομπέ, ε, κατά 8% επιβαρύνουν τι εκπομπέ ε, θερμοκηπίου. Ο Καναδάς έχει τα καλύτερα αποτελέσματα μέχρι τώρα. Έχουν φτάσει στους 18 ορόφους και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα, στήσει, θα κτίσει ένα κτίριο 22 ορόφων που θα είναι το πιο ψηλό ξύλινο κτίριο στον κόσμο. Στη Βιέννη θα χτιστεί αυτό. Αυτά είναι κτίρια τα οποία βοηθούν στη δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακος. Σας κάνω λοιπόν μια έκκληση να δώσετε κίνητρα για να ενθαρρυνθεί η κατασκευή ξύλινων κτηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση είναι κάποιο, κάπως περίεργη γιατί όσο περισσότερα δάση έχει μια χώρα τόσο λιγότερο ψηλά ξύλινα κτίρια έχει. Οι σκανδιναβικές χώρες που έχουν τεράστιους πόρους ε, όσον αφορά ε, την ε, υλοτομία δεν έχουν ξύλινα κτίρια και αυτό έχει σχέση με ε, τους οικοδομικούς κανονισμούς, ιδίως τα μέτρα προστασίας ενάντια της φωτιάς. Αν μπορείτε λοιπόν να βοηθήσετε σε αυτόν τον τομέα στο Λουλουσία θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη η συμβολή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπράνεν. Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο? Αν όχι, ολοκληρώνουμε εδώ το δεύτερο γύρο. Και δίνουμε το λόγο και πάλι στον Υπουργό για να μας απαντήσει. Thank you. Many complicated... Πολλά και περίπλοκα ζητήματα, αλλά θα καταβάλω κάθε προσπάθεια ε, για να απαντήσω στις ανησυχίες που άκουσα. Καταρχήν, η ερώτηση της κυρίας Σάιερ Πίρικ σε σχέση με μια ισορρόπηση της διατήρησης της ε, φύσης και των συμφερόντων των εμπλεκομένων. Συμφωνώ μαζί σας ότι για να είμαστε επιτυχείς ως προς τη διατήρηση της ε, φύσης θα πρέπει να εμπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι το ότι οι δράσεις μας είναι χρήσιμες. Υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να εμπλακούν όλοι στη διαδικασία αυτή και πρέπει να συζητήσουμε μαζί τους και τα, τις επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων και τις επιπτώσεις στις διάφορες βιομηχανίες. Και έτσι μόνο θα μπορέσουμε να τους εντάξουμε στο σχέδιό μας και να είμαστε επιτυχείς. Το Συμβούλιο ενέκρινε τις αποφάσεις του υποστηρίζοντας το νέο πρόγραμμα δράσης για τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εποπτεύσει αυτό το πλαίσιο εφαρμογής μαζί με όλα τα θεσμικά όργανα. Και γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει το πρόγραμμα δράσης και την προσέγγιση των ε, πολλαπλών εμπλεκομένων. Προς τον κύριο Πάρμια θα ήθελα να πω τα εξής. Ως προς τον διάλογο με τις βιομηχανίες, στη ΣΥΠΑ, προβλέπεται μία άτυπη σύνοδος των Υπουργών Περιβάλλοντος στο Ταλίν αυτή τη εβδομάδα και την Παρασκευή θα συζητήσουμε την κατάσταση πραγμάτων ως προς τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα και πιστεύω ότι θα έχουμε επικοδομητικές διαπραγματεύσεις και φυσικά θα τεθεί και το θέμα της συμμετοχής άλλων εμπλεκομένων φορέων στις ΗΠΑ. Και αυτό το θέμα θα είναι επιτάπητος και ελπίζω να φτάσουμε σε μια κοινή συμφωνία. Προς τον κύριο Φαρία θα ήθελα να απαντήσω τα εξής. Μίλησε για την ε, στρατηγική κατά των πλαστικών, κατά του πλαστικού. Το πλαστικό μας περιβάλλει στην καθημερινή μας ζωή και συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν δυσίωνες προβλέψεις. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό θα έχουμε ακόμα περισσότερο πλαστικό στους ε, ωκεανούς που θα πλήξουν ε, τους ωκεανούς και τα ψάρια. Άρα η στρατηγική καταπολέμηση των πλαστικών θα είναι χρήσιμη προς αυτή την κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της απαλήφης τους. Αναμένουμε τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας της Κομισιόν σε σχέση με την ε, στρατηγική κατά των πλαστικών, αλλά και το πακέτο αποβλήτων θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτόν. Επίσης, η κυρία Μάισνερ και εσείς υποβάλατε το ερώτημα για τους ωκεανούς γενικότερα και το ρόλο της Προεδρίας μας. Φυσικά θα συμμετάσχουμε σε στην διάσκεψη των ωκεανών στη Μάλτα και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί προσδίδουμε μεγαλύτερη, όλο και μεγαλύτερη σημασία στους ωκεανούς, κάτι το οποίο ε, πήγει αν λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις απειλές. Έχουμε και μια πολύ ευρία ακτογραμμή στη χώρα μας και ανησυχούμε ιδιαίτερα για τις εξελίξεις. Επίσης θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στον ε, βιώσιμο στόχο 14 Η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών του Ιουνίου βοήθησε για να προσδώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην κατάσταση των ωκεανών μας. Ο πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος της ε, Εστονίας, ο Μάρκο Πόμερανς, ε, ε, κατήχε τη θέση του Αντιπροέδρου σε αυτή τη διάσκεψη. Άρα θα συνεχίσουμε να είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι σε αυτό το ζήτημα. Προς τον κύριο θα ήθελα να πω τα εξής. Μιλήσατε για το Λουλουσιεφ, αλλαγή χρήσης και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι στη διαδικασία αυτή και φυσικά, όπως ήδη αναφέρθηκε σήμερα, οι θάλασσες αποτελούν ένα δύσκολο θέμα και έχουμε να λογοδοτήσουμε. Και φυσικά χρειάζεται καλύτερη χρήση και περισσότερη χρήση ξύλου και υποπροϊόντων ξύλου σε όλα τα κράτη-μέλη. για να λάβουμε απαντήσεις ως προς πολλαπλές ανησυχίες. Χαίρομαι διότι ε, αναφερθήκατε στα ξύλινα σπίτια γιατί και στη χώρα μου, στην Εστονία, είμαστε ιδιαίτερα επιτυχείς σε αυτό το τομέα. Είμαστε η επικεφαλής χώρα σε ε, εξαγωγές ξύλινων σπιτιών. Και Είμαστε πολύ επιτυχείς ως προς τις εξαγωγές ξύλου, αλλά θα έπρεπε να είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι και στην πατρίδα μου. Και ε, θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Γκούτελαντ για, ως προς την ερώτηση που υπέβαλε για το ETS τους διάφορους ε, τομείς μεταφορών. Κατανοώ την ανησυχία σας. Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν, υπάρχει ένα θέμα εδώ σε σχέση με τους διάφορους ε, τομείς μεταφορών και υπάρχει μεγάλη ανησυχία ως προς τις ανισότητες ε, μεταχείρισης των διαφόρων τομέων. Αυτό αφορά και τον τομέα της ε, αεροπλοείας, του σιδηροδρόμους, τις θαλάσσιες ε, μεταφορές, πέρα από τις οδικές και η λύση για τις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Και η συζήτηση θα πρέπει να γίνει στο Διεθνή Οργανισμό της Θάλασσας, στο IMO. Προς τον κύριο Λάινεν θα ήθελα να απαντήσω τα εξής. Ε, μιλήσατε για τους ε, πόρους χρηματοδότησης στη διατήρηση της φύσης. Θεωρώ ότι είναι ζωτικής ε, σημασίας και έχει μεγάλη σημασία και στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε ε, είναι να λάβουμε υπόψη και την προτεραιότητα της οικολογικής καινοτομίας για να βρούμε τις ε, καλύτερες λύσεις χρηματοδότησης ε, σχεδίων οικολογικής καινοτομίας για να ξεκινήσουν αυτά τα σχέδια και να υποστηρίξουμε και συναφή προγράμματα, τα οποία θα οδηγήσουν σε μεγάλες αλλαγές σε πολλαπλούς τομείς. Επίσης υποβλήθηκαν ερωτήσεις για το πακέτο ενέργειας και άλλα ζητήματα τα οποία εμπίπτουν στο, εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο συναδέλφων της Εστονικής Προεδρίας και θα επανέλθω με απαντήσεις γραπτός. Όταν έχω περισσότερες πληροφορίες από τους συναδέλφους και τις οποίες θα σας δώσω με χαρά γραπτός. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Uh, ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε, σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας Ελπίζω μαζί με τους συναδέλφους να μπορέσουμε να συνεργαστούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα ζητήματα που μας απασχολούν. Ευχαριστούμε πολύ, σας εύχομαι κάθε επιτυχία και εγώ προσβλέπω στη συνεργασία μας.